Κυρία Μπένοβα, επεξήγηση ψήφου. Prego. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Μπορείτε ίσως να χρησιμοποιήσετε το διπλανό. Δεν λειτουργεί κανένα. prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Παρακαλώ να ελέγξουν οι υπηρεσίες γιατί δεν λειτουργεί κανένα μικρόφωνο. Vuol riprovare, onorevole Benova? Cosa? Sì. Europa, Sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Γίνονται προσπάθειες επίλυσης αυτού του τεχνικού προβλήματος από τις υπηρεσίες μας. mi dispiace Λυπάμαι κυρία Μπένοβα, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα ανεξάρτητο της ε, βούλησης της Προεδρίας, πρέπει να περιμένετε. see. Wow. Okay, it's work. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Prihlásila som sa na vysvetlenie hlasovania. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα απλά να κάνω επεξήγηση ψήφου για την έκθεση πρωτοβουλίας Λέχνερ, διότι θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση. Σχετικά λοιπόν με την έκθεση ε, Λέχνα, αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολύ σύντομα να πω ότι είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία πολύ σημαντική. Τη συζητήσαμε χθε το βράδυ. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία προτείνει τη διασύνθεση των μητρών επιχειρήσεων ή ανάλογων μητρών των ε, νομικών προσώπων των κρατών μελών προκειμένου να έχουμε αξιόπιστες ε, και καλές πληροφορίες και και τα λοιπά και για τη δημιουργία μιας ε, μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου. Είναι απαραίτητη λοιπόν η συλλογή δεδομένων για κάθε νομικό πρόσωπο προκειμένου να καταστεί δυνατή διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου να ενισχυθεί η μια αγορά. Και θα πρέπει και με το e-justice βέβαια να γίνει και η απαραίτητη διασύνδεση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κυρία Μπένοβα, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που μείνατε και μέσα στο λεπτό που επιτρέπει ο χρόνος. Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε το έργο Dr. Ζιβάγκο, όπου η μπουρζουαζία και η ιστοκρατία απολαμβάνουν σαμπάνια μέσα στην ζεστή ατμόσφαιρα ενός εστιατορίου ενώ έξω διαδηλώνει ο κόσμος. Και σήμερα το πρωί ε, θυμήθηκα αυτή την κινηματογραφική ταινία γιατί το Ευρωβαρόμετρο μας δείχνει σε σφιγμομετρήσεις ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της. Αλλά ακούσαμε τον κύριο Φερχόφστα, τον κύριο Ντόλ και άλλους ότι αυτό συμβαίνει γιατί εμείς δεν κάνουμε αρκετά διότι θέλουν η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Και ακούσαμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής που λέει ότι φταίνε τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι η ανθρώπινη φύση που προσπαθεί να αποφύγει το να αυτοκατηγορείται για το ότι δεν είναι κανείς δημοφιλής. Αλλά δεν μπορούμε παρά να δούμε ότι αυτό είναι μια ένδειξη που έχει σχέση και με το ευρώ και με τις διασώσεις επιχειρήσεων ε, και ε, με τα κεφάλαια και με τον τρόπο με τον οποίο ε, απαξιώνουμε τα αποτελέσματα εκλογών. Και κλείνοντας με τα λόγια του Edmund Burke, θα ήθελα να πω ότι μπορεί λίγες ε, ακρίδες ε, να κρύβονται μέσα στο γρασίδι την ώρα που ε, λίγο πιο πέρα βόσκουν ήρεμα οι αγελάδες ενώ όλοι είναι κάτοικοι του ίδιου χωραφιού.

η συμφωνία με την Κορέα είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να ελέγξουμε και δεν μπορεί να δεσμεύεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πρόκειται για επιστροφές και μηδενικούς τελωνιακούς δασμούς από την Κορέα. Είναι ένα βήμα χωρίς προηγούμενο, απελευθέρωση της αγοράς που δεν φέρνει κάτι σε αντιστάθμισμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν υποστηρίζω τη συμφωνία με την Κορέα. Και υπάρχει και μια έκθεση η οποία προσπαθεί να ε, ρίξει φως σε όλα αυτά τα θέματα θέματα και η συμφωνία θα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί πριν την επικύρωσή της. Διαφορετικά υπονομεύουμε την ευρωπαϊκή αυτο... αυτοκινητοβιομηχανία. Χαίρομαι που αναβλήθηκε η ψηφοφορία. Volevo essere certo eh, che la prenotazione eh, θα ήθελα να είμαι σίγουρο, ότι έχει ε, σημειωθεί το όνομά μου για την έκθεση Μπίνευ και την έκθεση Βίνκλερ. Ξεκινήσατε με εκθέσεις οι οποίες ακολούθησαν τις δύο αυτές. Θα ήθελα να μάθω αν θα μου δώσετε το λόγο γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να είμαι εδώ. Σε αυτές τις εκθέσεις τις οποίες αναφέρατε δεν έχει υπάρξει συζήτηση και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχουν και επεξηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν επεξηγήσεις ψήφου γιατί δεν έχει υπάρξει συζήτηση και τροπολογίες. Για αυτές τις δύο, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος, δεν θα υπάρξουν επεξηγήσεις ψήφου. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μποβέ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπαρτολότσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σχετικά με τα εισοδήματα των Ευρωπαίων αγροτών, αν συγκριθούν με τα κέρδη της ε, βιομηχανίας που επεξεργάζεται τα τρόφιμα, οδηγούμεθα στην περιφερειοποίηση την οικονομική του γεωργικού τομέα και στη μείωση των δραστηριοτήτων των γεωργικών φυσικά. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η έκθεση την οποία συζητήσαμε σήμερα και για την οποία εκφράζω την υποστήριξή μου προτείνει συγκεκριμένα μέτρα κατά τομέα και νομοθετικές προτάσεις. Αυτά αφορούν όχι μόνο τα γεωργικά προϊόντα αλλά και την διασφάλιση προμήθειας πρώτων υλών για τον γεωργικό τομέα. Αυτό δεν είναι θέμα δικαιοσύνης μόνο για τους γεωργούς αλλά ενισχύει και την διαπραγματευτική τους ισχύ και αποτρέπει καταχρήσεις από πλευράς άλλων οικονομικών εταίρων. Είναι απαραίτητο να ληφθούν λοιπόν μέτρα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας. Ευχαριστώ κύριε Μπαρτολότσι. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα λάβαμε μια σωστή απόφαση, μια απόφαση καλή για τους αγρότες, καλή για τους καταναλωτές και καλή για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Το πιο σημαντικό σε αυτή την πρόταση πρωτοβουλία είναι το πολιτικό μήνυμα που δίνουμε. Ένα πολιτικό μήνυμα προ την αλυσίδα εφοδιασμού τη αγορά ότι όλοι και ιδίω οι αγρότε έχουν δικαίωμα για σωστή ανταμοιβή τη εργασία του. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όπω μέχρι τώρα. Δεν διαφωνώ να έχουμε σε σωστές τιμές τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να τηρούνται οι προϋποθέσεις ε, για την σωστή ενεργειακή αξία αυτών των ειδών που αγοράζουμε, γιατί όταν η ποιότητα αυτών των προϊόντων δεν είναι η σωστή, τότε κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα. Θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και ο ανταγωνισμό και όταν δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμό, θα πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτική και γι' αυτό η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Μαγκίνε. Ευχαριστώ. Να υποστηρίξω και εγώ την έκθεση Μποβέ και να συμφωνήσω με τα σχόλια του συναδέλφου ότι στέλνουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όσου ε, και όσου ασχολούνται με την πολιτική στην οικονομική αλυσίδα. Ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σοβαρό σε ό,τι αφορά ε, τη δουλειά του. Είχαμε μια συζήτηση για το περιεχόμενο τη έκθεση. Συμφωνούμε όλοι ότι οι αγρότε ε, δεν μπορούν πλέον να αφαιμάσονται και να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερε δυσκολίε. Καταλαβαίνουν πληρώνοντα το τίμημα ε, για, για τα προϊόντα αυτά τα οποία εμεί αγοράζουμε. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό, θα πρέπει να δούμε τους ε, που βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση, να δούμε τι γίνεται στον τομέα, τι κάνει η παγκόσμια οικονομία ε, για τους παραγωγούς τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει ένα σωστό νόμος περί ανταγωνισμού και ε, χαίρομαι που έλαβε τη δέουσα υποστήριξη αυτή η έκθεση γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να στηρίξουμε τα λόγια που ακούγονται τον τελευταίο χρόνο με πράξεις. Ρόιτοβα. για την έκθεση σε ό,τι αφορά τα δίκαια εισοδήματα και τους γεωργούς. Χαίρομαι πολύ που η Επιτροπή Γεωργίας ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα της βελτίωσης της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού, είδε τις διαφορές μεταξύ των χαμηλών τιμών ε, των γεωργών και των υψηλών τιμών πρέπει να καταβάλουν οι Θέλω να αναφέρω επίσης ότι είναι παράδεκτη η διάκριση και ο αθέμητος ανταγωνισμός που υφίστανται οι ε, γεωργοί των 12 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των επιδοτήσεων. Στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη, οι αγρότες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αγαθά όπως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα από την Τσεχία διότι προτιμώνται οι τα φθηνότερα προϊόντα από τις άλλες χώρες, τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ την κυρία Ροϊτόβα.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 Αυτή η έκθεση μιλά για τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να διασφαλίσουμε για τους αγρότες και είναι μια σημαντική έκθεση γιατί έχουν, ε, έχει ανέβει το κόστος παραγωγής και το κόστος αγοράς των προϊόντων και γι' αυτό πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις ε, επί των αγροτών και επί του εισοδήματός τους. Οι καταναλωτές ε, δεν θα πρέπει να είναι αυτοί που θα βγαίνουν χαμένοι. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν πάντοτε η προστασία της ποιότητας ζωής των αγροτών, αλλά δεν μπορούμε παράλληλα να διασφαλίζουμε ε, όλους τους στόχους. Θα πρέπει να βρεθεί και κάποια συμβιβαστική λύση. Θέλουμε να έχουμε νέους ε, που θα δουλεύουν στον αγροτικό τομέα, ενώ στη χώρα μου ε, πολλοί νέοι εγκαταλείπουν την αγροτική παραγωγή και γι' αυτό ίσως ε, χρειάζεται να δούμε το θέμα των ενισχύσεων που τους δίνουμε. Και εδώ υπησέρχονται και τα θέματα των κριτηρίων συνοχής. Εγώ υποστηρίζω την έκθεση αυτή και ιδίως Υποστηρίζω το ότι πρέπει να δούμε το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων εις βάρος των αγροτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στο σαν Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαρά μου υποστηρίζω την έκθεση αυτή. Ο τίτλος ε, τα λέει όλα. Δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα εισοδήματά τους δεν ήταν δίκαια και ευτυχώς κάνουμε τώρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση διότι θα πρέπει το κέρδος ε, να το μοιράζονται και η παραγωγή ε, και όλη η αλυσίδα μέχρι τη λιανική πόλη. πράγμα μέχρι τώρα δεν γινόταν. Δίνουμε λοιπόν το σωστό μήνυμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε μια σωστή κοινή αγροτική πολιτική για να εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του οικογενειακού αγροκτήματος και τη βιωσιμότητα της γεωργίας στο μέλλον. Κάναμε λοιπόν ένα σωστό βήμα, ένα πρώτο βήμα για σήμερα και ελπίζω στο μέλλον να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλη. Και περνάμε στην έκθεση Πόρτα. Δίνω το λόγο στην κυρία Ρωμάνα Τζόρνταν Σιτσέλη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 Και στην έκθεση αυτή ε, μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση. Η αλληλεγγύη για πολλούς είναι μια αφηρημένη έννοια. Υπάρχει όμως ένας μηχανισμός από τον οποίο πρέπει να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει επαρκώς ο μηχανισμός αυτός ε, και προσδοκώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει μια αναθεώρηση έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά την εξαρτησία αυτού, αυτών των κονδυλίων και θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο οι πόροι αυτοί θα διατίθενται επάπειρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να προωθήσει την απασχόληση και με διαφορετικά ε, μέσα θα πρέπει να φροντίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα προστατεύει εκείνου οι οποίοι δεν προσαρμόζονται στους, ε, στις συνθήκες της αγοράς που τροποποιούνται. Ευχαριστώ. Κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα. Ε, Σαν σκιώδη συζητήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, importante lavoro svolto in apertura, e soprattutto in collaborazione σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες θεωρώ ότι η έκθεση αυτή περιλαμβάνει σημαντικά σημεία για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Οι προτάσεις αυτές είναι συμβατές με αυτά τα οποία είδαμε στα πλαίσια της αξιολόγησης που κάναμε στις αρχές του 2010 στο εσωτερικό της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ανταποκρίνονται σε μια επιθυμία ε, επιτάχυνσης και απλούστευσης ταυτόχρονα των διαδικασιών. Στα πλαίσια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και του αυξανωμένου αριθμού αιτήσεων υποστήριξης από όλα τα κράτη-μέλη θα ήθελα να υπογραμμίσουμε στο εσωτερικό της έκθεσης την δυνατότητα διεύρυνσης μέχρι το 2013 της κάλυψης του ταμείου αυτού για απολυθέντες εργαζομένους λόγω της οικονομικής κρίσης. Ζητείτε λοιπόν από τα θεσμικά όργανα να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα και το ΦΕΔ νομίζω αποτελεί ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο στρέφεται προς τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει αγγλικά ο Πρόεδρος, την κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ θα πρέπει να φροντίσουμε να θυμόμαστε ότι αυτό το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να σταματήσουμε την απώλεια θέσεων εργασία και για να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Θα πρέπει να δίδονται 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίω για να επιτύχουμε του στόχου αυτού και θα πρέπει να φροντίσουμε να υλοποιούνται πραγματικά τα όσα ε, αναλαμβάνονται. Υπάρχουν νέα κράτη-μέλη που δεν έχουν υποβάλει αιτήματα για χρηματοδότηση. η Επιτροπή αποφάσισε να απλουστεύσει τη διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να συνεχιστεί. Όσον αφορά τις νέες χώρες όπου υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε τέτοιες μικρές επιχειρήσεις δεν εργάζονται πολλοί εργαζόμενοι, ακριβώς εκεί πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να βοηθήσει ακριβώς αυτούς τους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Σικιώσκη. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητήσαμε μια σημαντική έκθεση για τα δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες και τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που εξαρτάται και από το δρόμο που διανύουν τα προϊόντα, δηλαδή από το αγρόκτημα προς ε, τους καταναλωτές. Ε, είναι πολύπλοκη η γεωργική δραστηριότητα Και ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει και πολλά ο αγρότης ε, για τις συνθήκες και την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ των τιμών ε, των γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει να καταστήλουμε τις μονοπωλιακές δραστηριότητες από πλευράς αλλιανοπολιτών. Θα πρέπει τα, οι εθνικοί φορείς να παρακολουθούν την κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει απουσία ελέγχου. Υπάρχει κατακαιρματισμός και απομόνωση και έτσι η απώλεια των εισοδημάτων των αγροτών. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τσβίφκα. Ο κύριος Μπουρνογκολνής έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του συναδέλφου Τσβίφκα δείχνει μεγάλες γνώσεις και επεξεργασία και ε, των κοινωνικών νομοθετημάτων, της νομολογίας, ε, που γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές ε, χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Η έκθεση αυτή ένα μέρος του προβλήματος όμως μόνο επιλύει. Πρόκειται πάντως για ένα τομέα που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα είχε πλήρη νομιμοποίηση όχι δηλαδή τυποποίηση ε, του ουσιαστικού δικαίου, αλλά εναρμόνιση κάποιων κανόνων που αφορούν σύγκρουση νομοθεσιών για να δούμε ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο και εναρμόνιση κάποιων κανόνων σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση δικαίου, όπου πρέπει να δούμε ποιο δίκαιο θα εφαρμόζεται σε σχέση με τις συμβάσει, αν ε, κάποιο βρίσκεται σε ένα διαφορετικό χώρο, άλλη περιουσία, κινητά, περιουσιακά στοιχεία, σύμβαση των συμβαλόμενο είναι σε διαφορετικό μέρος κτλ. Όλα αυτά κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να επιλύονται με ένα ευρωπαϊκό κώδικα. Αν δεν υπάρχει αυτός ο κώδικας ευρωπαϊκού ιδιωτικού ε, δικαίου δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ σημαντικέ δυσκολίε που η έκθεση αυτή πολύ σωστά εν μέρη τουλάχιστον επιλύει. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το εξυπεκβάτουρ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μικολάσιτ. There is not. Δεν παρίσταται ο Κύριος Μικολάσιτ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρόιτομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους τάκτες της έκθεσης ότι μάλλον τη συντάκτρια τη ε, έκθεση, ότι υπάρχουν αρνητικέ διακρίσει σε βάρο γυναικών που ανήκουν σε ομάδε εθνικών μειωτοτήτων. Θα πρέπει να κάνουμε το πάνω στο να βελτιωθεί η κατάστασή του, σε ό,τι αφορά την πρόσβασή του, την εκπαίδευση, στην ε, υγειονομική περίθαλψη, την αγορά εργασία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις στατιστικές, ε, τα στατιστικά στοιχεία ανά εθνοτική μειονότητα, πρέπει να πω ότι η νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύει κάτι τέτοιο. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει κατά πόσον θα μπορούσε ε, να γίνει αυτή η συλλογή στατιστικών στοιχείων χωρί να καταπατώνται οι νομοθεσίε. Μπορούν να γίνουν ε, τέτοιε αναλύσει. Η συντάκτρια και το κοινοβούλιο έχουν υπόψη ότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι είμαι υπέρ τη έκθεση. voorzitter. Κύριε Σούλιφ Κλέης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της έκθεση, Παρβάνοβα. Η κοινωνική ένταξη των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες είναι μια έκθεση για την οποία ψήφισα κατά, διότι πιστεύω ότι είναι αντιπαραγωγικό το να κάνουμε τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις. Αποφεύγουμε να αναφέρουμε το Ισλάμ και είναι γελίο. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η διακριτική μεταχείριση της οποίας ε, είναι θύμα οι γυναίκες ε, ξεκινά από την ίδια την κοινότητα κυρίως για θρησκευτικού λόγους. Φοβόμαστε όμως να το αναφέρουμε και να θέσουμε το δάκτυλο επί του τύπου των ήλων ε, για μια πραγματικότητα αυτά τα οποία προσωπεύει το Ισλάμ δεν επιτρέπουν ε, την ένταξη στην ευρωπαϊκή μας κοινωνία. Όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρνείται να το αναγνωρίσει, δεν θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την ένταξη των γυναικών που προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες, εάν δείξουμε υπερβολική ανοχή. Ευχαριστώ. Έκθεση Πιετικάινεν και δίνω το λόγο στον κύριο Καλινόσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι ουσιαστικά άχρηστοι σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι έχουν σημαντική μεταδοτική εμπειρία όσον αφορά τη μεταδοτικότητα και οι γυναίκες επίσης είναι πολύ χρήσιμες παρά τις ε, διακρίσεις οι οποίες πάντα υπάρχουν και γι' αυτό άλλωστε και πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες από αυτά τα προβλήματα όπως είναι η φτώχεια ή η διαφορά στους μισθούς. Αυτά τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα εμφανή στην Ήπεθρο. Χαίρομαι πολύ λοιπόν ε, που εγκρίναμε αυτό το ψήφισμα γιατί μας επενθυμίζει τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μας κινητοποιεί να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μακκίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω την έκθεση αυτή και θα ήθελα ιδιαίτερα να επιστήσω την προσοχή σε τρεις πολύ σημαντικές κατεμέ παραγράφους για να μην ε, βάζουμε τους ανθρώπους σε κάποια ιδρύματα μέρη ή να τους φροντίζουμε στο σπίτι. 17, 19 και 25 είναι παραγράφοι πολύ ενθαρρυντικές προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά τη μέρημνα των ηλικιωμένων που θα βασίζεται στα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να ζουν ανεξάρτητα ηλικιωμένοι στο σπίτι τους. Πρέπει να υπάρχει σχετική υποστήριξη και θα πρέπει να υπάρχει κερδοσκοπία σε βάρο ε, των ηλικιωμένων ε, που θα περνούν ε, στον τομέα τη ιδιωτική μέρημνα. Παράγραφο 13 για τη συμφιλίωση εργασία και μέρημνα. Θέλω να πω ότι και εδώ και σε πολλά κοινοβούλια και στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα γίνονται προσπάθειε για την. θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες συμφιλίωση τη πολιτική εργασία, του πολιτικού έργου με την μέρημνα, γιατί υπάρχουν κάποιοι ε, πολιτικοί οι οποίοι έχουν και ρόλο φροντιστή και αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ερμήνια Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ψήφισα υπέρ της εκθέσεως αυτής γιατί περιλαμβάνει την επιβεβαίωση κάποιων βασικών για μένα αρχών. Η γύρανση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αρνητικό τρόπο, είναι ένα στοιχείο πλούτου για την κοινωνία μας. Οι οικονομικές κρίσεις φυσικά επηρεάζουν άμεσα τις γυναίκες και ιδιαίτερα τις γυναίκες μιας κάποιας ηλικίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών των ηλικιωμένων, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες υποφέρουν από την έλλειψη οικονομικών μέσων, ενώ ταυτόχρονα είναι τα θεμέλια, θα έλεγα, του λεγόμενου welfare. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τις μελέτες έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην προχωρημένη ηλικία που φυσικά είναι καρπός των διακρίσεων που έχουν υποστεί οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου της ζωής τους. Με αυτό το ψήφισμα ζητούνται τρία βασικά πράγματα θα έλεγα. Ένας μεχανισμός ο οποίος δίνει την δυνατότητα στη σώρευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ζητάμε να ληφθεί υπόψη η διάσταση της διαφοράς φύλου στα πλαίσια της ε, ε, ηλικίας συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα να καλυφθεί το πρόβλημα που υπάρχει στον τομέα της πρόνοιας αντιμετωπίζεται σοβαρό θέμα εδώ ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ιταλία και όπου τα εθνικά συστήματα δεν είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ευχαριστώ κυρία Ματσόνη. Και Λία Ρόιτοβα έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Γιατί η πρόταση λέγει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και των ομοφιλοφίλων. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά από ό,τι οι υπόλοιπε ας πούμε γυναίκες αυτούς, αυτής της κατηγορίας. οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα και τα εισοδήματά τους είναι χαμηλότερα γιατί φροντίζουν την οικογένειά τους. Αλλά αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Σον Κέλλη. Υποστήριξα και εγώ την έκθεση αυτή. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε μέρος στη συζήτηση χθε και ζήτησα να... Δεν πήρα το λόγο όμως γιατί θεωρώ ότι ο τίτλος της έκθεσης αυτής πιετικά είναι δεν ήταν ο πιο σωστός. Αντί να μιλήσουμε για τη γύρανση των γυναικών στην κοινωνία, μιλήσαμε για τη θέση των γυναικών σε μια γυράσκουσα κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή για τον ρόλο και των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία στα πλαίσια της προχωρημένης ηλικία και αυτό έχει άμεση σχέση και επιπτώσεις στον τομέα της οικονομίας και τον δημοσιονομικό. Η γυράσκουσα σε εισαγωγικά κοινωνία θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργεί και μέσα από τον προϋπολογισμό. Έκθεση Λόκερ Γκάρντα. Ο κύριος Μαστέλα έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την έκθεση Λόκεργαρτ γιατί θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για την κατανομή των σχέσεων και των ευθυνών και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει την αντιπροσωπευτικότητα της δημοκρατικής μας ε, μεθόδου. Το λέγω αυτό επίσης γιατί θέλω να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Ευρωπαίων στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Διαπίστωσα όμως ότι και στις τελευταίες ευρωεκλογές υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αποχή, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για τις διάφορες πολιτικές και τα θέματα και θεωρούν ότι τα όργανα τα ευρωπαϊκά είναι μακριά από αυτούς. Σύμφωνα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινοτική μέθοδο, θα πρέπει εμείς αυτήν την απόσταση που νιώθει ο πολίτης να βοηθήσουμε να την ξεπεράσουμε και να υπάρχει δωρεάν και εύκολη πρόσβαση, πρόσβαση σε όλες τις πηγές, ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης. θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις κοινωνικές και τις εθνικές αρχές που και αυτές να συμπληρώνουν την σωστή ενημέρωση και ο, ο Ευρωπαίος πολίτης να είναι πιο σωστά ενημερωμένος για ό,τι αφορά την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Μαστέλα. Ο κύριος Λόκεγκάρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι είναι θετικό το ότι έγινε δεικτή η έκθεση για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία. Νομίζω ότι μαζί με το αντίστοιχο ψήφισμα το νομοθετικό μας ε, δίνουν έναν σωστό τρόπο για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Υπήρξαν αρκετοί συμβιβασμοί βέβαια. Ε, θα ήθελα οι συμβιβασμοί αυτοί να γίνουν δεκτοί από όλους ε, τους εμπλεκομένους. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει εκφράζω την βαρέσκειά μου για τη συζήτηση που προηγήθηκε και ελπίζω ότι οι προτάσεις από εδώ και πέρα να γίνουν πραγματικότητα. Ε, I give κύριε Λόκερκαρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή με χαρά γιατί είμαι τέος δημοσιογράφος και γνωρίζω όλες τις πλευρές αυτού του θέματος και σαν δημοσιογράφος και σαν πολιτικός. Δεν πρέπει να ταυτίζουμε βέβαια την ενημέρωση με τη δημοσιογραφία και ταυτόχρονα η οικονομική κρίση ε, θέτει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων εκτός δουλειάς. Αυτό έγινε και σε μεγάλες εφημερίδες και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς υπάρχει πίεση για απολύσεις. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πτώση στην ποιότητα των, της ενημέρωσης γιατί δεν θα υπάρχει χρόνος και άνθρωποι για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει και εις βάρος της ευρωπαϊκής μορφής ενημέρωσης γιατί μπορεί να καλύπτονται ορισμένα τοπικά θέματα αλλά όχι τα ευρωπαϊκά θέματα ενώ θα πρέπει και τα ευρωπαϊκά να γίνονται γνωστά. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Βλάσσακ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, το θετικό της έκθεσης είναι ότι αναγνωρίζει επανειλημμένως ε, το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και τονίζει και τη σημασία της αρχής της επικουρικότητας. Συμπεριλαμβάνει επίσης προτάσεις για την αύξηση της διαφάνειας, της δημοσιοποίησης των πληροφοριών, διευκολύνοντας το έργο των δημοσιογράφων βέβαια. Απ' την άλλη πλευρά συμπεριλαμβάνει και κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα. Παραδείγματο χάρη προτείνει να υπάρξει ε, μια ομάδα ανταποκριτών που θα καλύπτουν ε, τα ευρωπαϊκά ζητήματα με πιο μορφωτικό ή παιδευτικό, αν θέλετε, χαρακτήρα και λέει επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εξειδικευμένο γραφείο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα σε κάθε χώρα που θα πρέπει να εξηγεί τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνει ταυτόχρονα τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωκοινοβουλίου να έχουν ε, μεγαλύτερο προπολογισμό. Νομίζω ότι καλύτερα αποτελέσματα θα επιτυγχάνονταν με πιο αποτελεσματικέ μεθόδου και όχι με την αύξηση του προπολογισμού. Γι' αυτό καταψήφισα. Ευχαριστώ. Είναι Σπάιντεφ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο θεωρώ θετικό είναι ότι στην έκθεση αυτή υπενθυμίζεται η ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι σημαίνει. Αυτό είναι η βάση της Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ευθύ, τις ευθύνες μας. Ε, διαθέτουμε πολλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γραφεία πληροφοριών ε, των κρατών μελών θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι μέχρι τώρα. Επιμένω στο γεγονός ότι η ροή πληροφοριών προς τα γραφεία πληροφοριών θα πρέπει να ελέγχονται. Από και προς μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους πόρους που διατίθενται στα γραφεία πληροφοριών. Χαίρομαι πολύ που γίνεται και η θετική αξιολόγηση του Euronews. Εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι το κανάλι αυτό που εκπέμπει σε όλες τις επίσημες χώρες είναι κάτι πολύ θετικό. Στη Λετωνία δεν μπορούμε παρά μόνο ρωσικά να ακούσουμε το Euronews. Δεν υπάρχει στα λετωνικά. Και αυτό με λυπεί προτείνω να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δώσει τη δυνατότητα τα mass media των διαφόρων χωρών να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και ανεξάρτητα, ιδίω όταν δεν υπάρχει στη χώρα η απαραίτητη πολιτική βούληση για την εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Thank you, President. Uh, this report and Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα για τα νέα μέσα ενημέρωση και τη δημοσιογραφία πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα νέα μέσα τροποποιούν και τη δημοσιογραφία και είναι σαν ευσεβή πόθη από πλευρά των Ευρωβουλευτών σχετικά με την χειραγώγηση του πόσο αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εγώ πιστεύω στην ελευθερία της έκφρασης και στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία και όχι στη χειραγώγηση της δημοσιογραφίας ε, για να καλύπτονται τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προάγουμε το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό είναι προπαγάνδα χάσαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τρόπους ε, δημοκρατικής ε, παρέμβασης στα μέσα και στην άσκηση δημοσιογραφίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας. Θα ξαναρχίσουμε στις 3.